οποίες ε, έχουν ε, υποβάλει κάποια διευθυντικά σε πέντε κείμενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το 231 θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά αυτά εκτός και αν υπάρχει ένταση μέσα, μέσα στις 24 ώρες και τα έχετε λοιπόν τα διορθωτικά αυτά στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας θα δημοσιευθούν και στα πρακτικά της συνεδρίασης μετά την διακοπή της, συνόδου τον Ιούλιο σύμφωνα με το άρθρο 78 μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου υπέγραψα 8 νομοθετικά κείμενα σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία.